Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους των ε, Πρασίνων Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, κυρία Σκοτ Κάτω. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στην προηγούμενη θητεία εκδώσαμε 15 ψηφίσματα για τη Βενεζουέλα και δεν είμαι πεπισμένη ότι οι πρόταση αυτέ είχαν σε στόχο να επιλύσουν την κρίση προ όφελο των περισσότερων Βενεζολάνων, αλλά να ενισχύσουν κάποιε φωνέ συγκεκριμένες και ε, από την άλλη λησμονούμε κάποιες άλλες φωνές και άλλα προβλήματα από τη Λατινική Αμερική που οδηγούν τώρα σε νέες μεταναστεύσεις και νέα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πραξικόπημα του Γουαϊδό προφανώς απέτυχε και μάλιστα παρατηρώ κυρία Μπογκερίνου, ότι καν το αναφέρατε στην ομιλία σας σήμερα. Από το τελευταίο ψήφισμα μας έχουμε σαν αποτελέσμα ότι η Μισελ Μπασλέ επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα, καταδίκασε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, αλλά κανείς δεν προχώρησε στην υλοποίηση της προ... των συμφωνηθέντων στο Μπαρμπέιντος. Πρωτοβουλία αξιέπαινη πράγματι. Ελπίζουμε όμως ότι μπορεί να καταλήξουμε σε μια διαμεσολάβηση για λύση, σε μια δημοκρατική διαδικασία την οποία να μπορούν να ενστερνιστούν όλοι οι Βελεζολάνοι και αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει το σώμα. Ευχαριστώ. Ομάδα Ταυτότητα Δημοκρατία, κύριος Ολιβιέ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Βενεζουέλα είναι πρώτα απ' όλα ανθρώπινη τραγωδία και η επιβεβαίωση ταυτόχρονα και του πόσο βλαβερές μπορεί να είναι κάποιες ε, κολεκτιβιστικές θεωρήσεις και προσδοκίες. Βλέπουμε ένα διπλό σφάλμα εμείς εδώ και την ε, έκφραση μιας ε, υποταγής, δηλαδή την τυφλή παρακολούθηση από πλευράς του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου Γουαϊντό των ε, επιταγών του Προέδρου Τραμπ. Τι άλλο λοιπόν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το να μετατρέπεται τελικά σε έναν μπαϊρακτάρι της ε, αστερόεσας. Αλλά και βλέπουμε ε, το άλλο λάθος την παρέμβαση, σκληρή παρέμβαση σε μια εσωτερική κρίση που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εμφύλιο πόλεμο. Η Ιταλία διατήρησε στάση αποστάσεων με όραμα, με διορατικότητα, κράτησε στάση αποστάσεων, πράγμα το οποίο δεν έπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τώρα βρίσκεται στη δύσκολη κατάσταση να διεκδικεί το ρόλο του διαμεσολαβητή. Ελπίζω αυτό το κακό ε, προηγούμενο αυτή η μεγάλη τροεγωδία να, μας να είναι ένα μάθημα για όλους. Μας ευχαριστώ κυρία Φωτσίκα εκ μέρους των στηρητικών μεταρρυθμιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Το 2017 δώσαμε το βραβείο Σαχάροφ στην αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα. Δυστυχώ, το καθεστώς Μαδούρο εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρό ακόμα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μαζικέ παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκφοβισμό της δημοκρατικής αντιπολίτευσης και μαζικέ συλλήψει. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα ε, και όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε τον υπερπληθωρισμό, τις ασθένειες, την έλλειψη βασικών αγαθών και ιδιαίτερα και τα βάσανα των ηλικιωμένων και των παιδιών σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει η μεταναστευτική κρίση που επηρεάζει αρνητικά και συνολικά την ε, περιφέρεια, την περιοχή την ευρύτερα. Όμως υπάρχει ελπίδα σε ό,τι αφορά τι διπλωματικέ προσπάθειες. χαιρετίζω την ε, ε, πρωτοβουλία των Ίσων Παρμπέιντος ε, που, ε, της οποίας ηγεί την Νορβηγία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Νοτικής Αριστεράς, ο κύριος Πινέντα Μαρίν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα Καταλανό πολιτικό του προηγούμενου ένα έλεγε ότι στην πολιτική μπορεί να κάνει ποιο, ό,τι θέλει εκτό από το γελίο. Αυτό που θα κάνει αυτό το κοινοβούλιο, αν εγκρίνει αύριο το νιωστό ψήφισμα για τη Βενεζουέλα, το κοινοβούλιο με τον Αγιντόνιο Ταγιάννη αναγνώρισε τον Γουαϊδοϊδό ω πρόεδρο μια χώρα που, αν και δεν σας αρέσει, έχει εκλεγμένο πρόεδρο ε, και απέτυχε το πραξικόπημα και ακριβώς όταν ο Γκοϊδό ε, πηγαίνει στην στροπέζη του διαλογού στον Περβάντος, ε, επιστρέφουν οι πιέσεις εσείς, συνεχίζετε με το χαρτί για να ρίξετε το Μαδούρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σεβαστεί όμως το διεθνές δίκαιο, την μη παρέμβαση στην εσωτερικά των λαών. Λέτε ότι ανησυχείτε για το λαό τη Βενεζουέλας, όμω απαιτείτε μέτρα που θα προκαλέσουν περισσότερα δεινά. Κυρία Μογκερίνη, σταματήστε να απειλείτε με κυρώσει και να ζητήσετε διάλογο και με τριοπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιλέξει και να προωθήσει το διάλογο και να αφήσει το λαό τη Βενεζουέλας να αποφασίσει για το μέλλον του. Θα πρέπει λοιπόν να δράσει δημοκρατικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ. Παρακαλώ κύριος Ρούλαντ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε Καστάλτο, ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση σήμερα στη Βενεζουέλα είναι παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν η σολιστική ιδεολογία επιδιώκεται μέχρι της ακραίας της έκφρασης και αυτό που με ανησυχεί ιδιαιτέρως μίστερα από τα όσα άκουσα από τους ευρωβουλευτές της αριστεράς είναι ότι θεωρούν πως πιο κεντρική οργάνωση ε, ρυθμίσεις και τα λοιπά μπορούν να οδηγήσουν σε μια ε, ουτοπική υπέροχη κοινωνία. Όχι, αυτό είναι αυταπάτη. Περισσότερη οικονομική ελευθερία είναι αυτό το οποίο μπορεί να επιτύχει την ε, καλή λειτουργία της κοινωνίας. Ο Φρέντρικ Χάιεκ, αυστριακός ε, οικονομολόγος είχε πει ότι ο κομμουνισμός θα οδηγήσει, ο σοσιαλισμός θα οδηγήσει στην υποδούλωση. Αυτό βλέπουμε να συμβαίνει και στη Βενεζουέλα όπου δεν έχουν ούτε φαγητό ούτε φάρμακα, όπου έχουν ε, πληθωρισμό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο της 100 και αναμένεται να, περισταλεί ακόμα περισσότερο η οικονομία του τα επόμενα χρόνια δεν βοηθάτε με αυτά που κάνετε τον θαραλέο Χουάν Γουάιντο, τον γενναίο αυτόν ηγέτη της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ πολύ και υπάρχει μια μπλε κάρτα αν τη δέχεστε κύριε Ρόλαντ. Ο κύριος Χόρουντ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ για τις σαφείς τοποθετήσεις του τον ε, κύριο Ρόλαντ, αλλά ε, πώς θα πείσετε την είπατε εκπρόσωπο όταν θα προχωρήσουμε στο Brexit. Απάντηση. Μα με πολυμερείς διαπραγματεύσεις την απάντηση του κύριου da... Ευχαριστώ και για την ερώτηση και για την απάντηση. Και τώρα Λόπες Χίλ, ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Μογκερίνη, ως ε, πολίτη τη Βενεζουέλη, αλλά ε, και Ισπανό, ε, σα μιλώ πολύ συγκινημένος. Είπατε εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, η κυρία Μπατσελέ, παρουσίασε την έκθεση τη για την παραβίαση των δικαιωμάτων των Βενεζολάνων ε, και μίλησε για βασανιστήρια, για διώξεις, ε, για ε, δολοφονίες σαν κρατική πολιτική και όπως το κατήγγειλε και εδώ η Δημοκρατική Αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο του 2017 κέρδισε το βραβείο Σαχάρος η νόμιμη Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας υποστηρίζει ότι πρέπει με το διάλογο να επιλύθει αυτή η κρίση ως συντονιστής Υποεπιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ευχαριστώ την δέσμευση για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος προκειμένου να υπάρχουν ελεύθερες και διαφανείς προεδρικές εκλογές υπό ε, την διεθνή, ε, διεθνείς εκλογικούς Στι 28 Μαρτίου αυτό το κοινοβούλιο ενέκρινε ένα έγγραφο που ε, ουσιαστικά προκρίνει την συνεργασία της ομάδας επαφής με την ομάδα της Λίμας. Αυτή είναι η μόνη οδός για τον εκδημοκρατισμό της Βενεζουέλα. Ζητώ από όλε τις δημοκρατικές πολιτικές ομάδες να υποστηρίξουν αυτό το ψήφισμα. Ο μόνος σκοπός είναι να πετύχουμε να σταματήσουν οι διώξεις ε, και οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η άσκηση βίας αλλά και μαζική έξοδος ε, των πολιτών της Βενεζουέλας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν πρόκειται να ξεπεράσετε το χρόνο σας, θα πρέπει να ζητάτε από τις ομάδες σας να σας δίνουν περισσότερο χρόνο. Μην μου δυσκολεύετε το έργο. Σάντος, ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρία η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα συνεχίζει να σοκάρει όλου του διεθνεί παρατηρητέ. Η έκθεση των ΗΕ μα δείχνει ότι η κατάσταση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλαπλασιέζεται και αγνοούνται οι κανόνε του κράτου δικαίου και οι συνθήκε διαβίωση του πληθυσμού είναι όλο και πιο δύσκολε. και κανείς δεν μπορεί να ε, ανέχεται αυτή την κατάσταση. Όμως, α είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει καμία λύση για τη χώρα ε, που να μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους που μένουν εκεί, που να μην περνά από το διάλογο και από τη διεθνή διαμεσολάβηση, προκειμένου να υπάρξει ειρηνική επίλυση της κρίσης. Ε, το έργο του Contact Group έχει ε, αποτελέσματα που αναγνωρίζονται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίζει να ασκεί πίεση για να ξαναυπάρξει θεσμική ισορροπία και για να εφαρμοστούν οι απαραίτητες αλλαγές για την υλοποίηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών ανοιχτών στη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων και με εγγύησης διεθνής παρακολούθησης, διεθνής παρατήρησης. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Και τώρα... Η κυρία Ραφαέλα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι πραγματικά προβληματική και θλίβει εκατομμύρια κόσμου. Τέσσερα εκατομμύρια έχουν φύγει από τη Βενεζουέλα. Σημαίνει ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κρίση εκτοπιστέντων στον κόσμο μετά τη Συρία. Εμείς όμως οι Ευρωπαίοι δεν ακολουθούμε τους ε, κανόνες που έχουμε θεσπίσει, αλλά και την ηθική μας υποχρέωση να υποδεχθούμε αυτούς που αιτούνται προστασίας. Και στην αρχή της χρονιάς πήγα ε, στο καρεβικό τμήμα της, ε, του Βασιλείου των Κατοχωρών. Τα είδα λοιπόν η διεισόμαση και είδα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί σε ό,τι αφορά την υποδοχή των προσφύγων. Ήδη λοιπόν στα νησιά αυτά πάνω από το 10% του πληθυσμού είναι πρόσφυγες. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει την απαραίτητη συνδρομή και όλα τα κατάλληλα μέσα. Πρέπει να κατανείμουμε πόρους, να αποστείλουμε εμπειρογνώμονες από το ΕΑΖΟ και περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέρτς για ένα λεπτό. Χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Μογκερίνη που πετύχαμε ένα ψήφισμα και ελπίζω να ψηφιστεί από ευρεία πλειοψηφία σε αυτό το νέο κοινοβούλιο προκειμένου να καταδείξουμε την τραγωδία που λαμβάνει η χώρα στη Βενεζουέλα εδώ και πολλά χρόνια και με πάρα πολύ απάθεια από την πλευρά πολλών. Ε, ακριβώς ε, έχετε αυτό το λυπηρό ρόλο που ε, παίξαμε. Δηλαδή υπήρξαν ε, στιγμές όπου θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν τα δεινά των Βενεζολάνων. Εδώ δεν μιλάμε ακριβώς ε, για μια ιδεολογική δικτατορία, αλλά μιλάμε για μια ομάδα εγκληματιών που προστατεύεται από ε, ένα κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στην Κούβα, στην Αβάνα και υπήρξε υπερβολική προστασία από αυτό το κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω και τη διάρκεια τη συζητητή σα. Η Κούβα είναι ένοχη για το τι έχει συμβεί στη Βενεζουέλα και δεν έχουν υποθεί τα πράγματα επαρκώ. Θα πρέπει να απειληθούν οι εγκληματίε στη Βενεζουέλα γιατί ε, διαφορετικά δεν θα κινηθούν οι διαπραγματεύσει ε, που θα λάβουν χώρα τώρα και θα πρέπει να υπάρχει επιλή για την επιβολή κυρώσεων ή οτιδήποτε άλλο σκεφτείτε είναι απαραίτητη όμως. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κούλογλου, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ε, Καλησπέρα κυρία Μογκερίνη. Ένα πολύ σαφές ερώτημα θέλω να σας θέσω. Πρόσφατα υπήρξε απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Βενεζουέλα. Γιατί δεν το έχετε καταδικάσει. Είστε υπέρ ορισμένων στρατιωτικών πραξικοπημάτων ή δικτατοριών. Γιατί όχι. Το δεύτερο ερώτημα. Πλέον υπάρχει κάποια πρόοδος πραγματευτική υπό την αιγίδα της Νορβηγίας. Γιατί υπάρχει μια τόσο επιθετική στάση και ψήφισμα. Γιατί δεν δίνεται σε αυτό το διάλογο μία ευκαιρία. Γιατί ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Και το τρίτο ερώτημα που έχω. Εάν ένας Γκουαϊδό εμφανιστεί σε άλλη χώρα, όπου έχουμε πολύ σοβαρές ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, που έχουμε ακόμα και ε, ανθρώπους που διαμελίζονται. Αν εμφανιστεί λοιπόν εκεί ένας ε, Γουαϊδό και εμφανιστεί ως ε, προστάτης ε, της δημοκρατίας, εκεί θα τον αναγνωρίζατε. Όχι. Α είμαστε ειλικρινεί λοιπόν, γιατί ε, στην Σαουδική Αραβία τα πετρέλα είναι ασφαλή, ενώ στη Βενεζουέλα όχι. Ευχαριστώ. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Ιβαν Σίντσιτς να λάβει το λόγο. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Ζήτησα το λόγο προκειμένου να μιλήσω κατά των στρατιωτικών εξοπλισμών υπέρ της ειρήνης, υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης της κατάστασης στη Βενεζουέλα. Μπορούμε να μιλούμε για, τα, για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, ναι. Γιατί όμως δεν γίνεται λόγος καθόλου για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Σαουδική Αραβία. Εκεί το κράτος ελέγχει τις ε, πετρελαϊκές πηγές και έτσι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ανθρώπινα δικαιώματα ούτε για τις γυναίκες συζητούμε ούτε ψηφίσματα εκδίδουμε για τη Σαουδική Αραβία και ρωτάμε από πού απορρέει αυτή η υποκρισία και πόσο θα κρατήσει. Θα ήθελα επίσης να στραφώ κατά του ιμπεριαλισμού των Ηνωμένων Πολιτειών είτε την εξουσία κρατούν δημοκράτες είτε ρεπουμπλικανοί, η ίδια εμπειριαλιστική πολιτική αναπτύσσεται σε σχέση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και δεν είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένε Πολιτείε παρεμβαίνουν στα εσωτερικά κράτους της Λατινικής Αμερικής. Πρέπει λοιπόν να καταδικάσουμε κάθε δικτατορία και να βοηθήσουμε τη Βενεζουέλα να αγωνιστεί και να σταθεί στα πόδια της κατά του υπεριαλισμού. Ευχαριστώ, Μίλαν, μόνο ένα λεπτό. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι όλο ένα και πιο δραματική. Το καθεστώς Μαδούρο, όπως είδαμε και από την έκθεση Μπατσελέ, παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες. Ουσιαστικά όλοι το ξέραμε και η δολοφονία ε, του καπιτάνιου Κώστα είναι πρόσφατη απόδειξη. Πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει καθυστέρηση, πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, να υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση και να υλοποιηθούν ελεύθερες προεδρικέ εκλογές. Ε, το νέο τραπέζι διαλόγου που προωθείται από την Ερβηγία θα πρέπει να παρουσιάσει σύντομα αποτελέσματα και να μην χρησιμοποιηθεί από το Μαδουρό για να κερδίσει χρόνο όπω συνέβη σε άλλες περιπτώσεις διαλόγου. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε μια πιο αποφασιστική στάση του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο προώθησε την ε, άμεση αναγνώριση του πριν κάποιου μήνε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί στενά με την ομάδα τη Λίμας ε, και με την πλειοψηφία τη διεθνού κοινότητα για να θέσει τέλο σε αυτόν τον τραγικό εφιάλτη που ζουν οι Βενεζολάνοι. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γουόρτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. The humanitarian... Η ανθρωπιστική, πολιτική και οικονομική κρίση στη Βενεζουέλα απαιτεί κατεπίγουσα ανταπόκριση. Η πρόσφατη έκθεση τη Υπόθεση Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, γιατί σκιαγραφεί μια πολύ ε, δύσκολη εικόνα ε, τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βενεζουέλα. Και το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα μπορεί να λυθεί μόνο μέσω μια διαπραγμάτευση που θα περιλαμβάνει όλες, ε, όλα τα τμήματα και τι κατηγορίε τη ε, κοινωνία. Πρέπει να συμμετάσχουν και οι μειονότητε, οι νέοι, οι γυναίκε, γιατί ε, έχουν στα χέρια του το κλειδί τη συμπεριληπτικής ειρήνης. Ελπίζω έτσι να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση μέσω της ε, ε, διαδικασίας συμφιλίωσης ε, που διοργανώνει η Νορβηγία. Και εμεί θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτέ τι συνομιλίε και να αντιταχθούμε σε οποιαδήποτε επιθετική λύση. Ο πόλεμο δεν είναι η λύση. Το μέλλον τη Βενεζουέλα δεν θα πρέπει να βασιστεί στη χρήση τη βία. Και οι συνομιλίε θα πρέπει να είναι επικοδομητικέ. Γι' αυτό καλό όλα τα μέρη να συνεχίσουν να εργάζονται θετικά προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών με παρουσία διεθνών παρατηρητών. Και υποστηρίζω απόλυτα ε, και το contact group και τα αιτήματά του, ε, μεταξύ άλλων και την ε, αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Κάρλο Φιντάντσα, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρετε κυρία Μογκερίνη. Έχει έρθει και η ώρα για τους απολογισμούς της δικής σας θητείας πέντε χρόνων και είναι αρνητικός για μας τουλάχιστον. Στη Βενεζουέλα όμως ξέρουμε ότι έκανε σημαντικές προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπούμαστε που πριν από μερικούς μήνες δεν μπόρεσε το Συμβουλίο να καταλήξει σε ένα ψήφισμα, σε ανακοίνωση που να υποστηρίζει τον ε, νόμιμο ε, ηγέτη τον Χουάν Γουαϊντό ακριβώς επειδή δική μου η χώρα η Ιταλία δεν θέλησε να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή έχουμε να κάνουμε με μεγάλη τραγωδία έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια μετανάστες γνήσιους μάλλον πρόσφυγες που αναζητούν βοήθεια δεν έχουν ε, όμως ε, το Ρομπέρτο Σαβιάνο να τους υποστηρίζει και έτσι κανείς δεν τους ξέρει. Είναι γνήσιοι πρόσφυγες όμως και πρέπει να αναπτυχθούν οι δυνάμεις μέσω και των διπλωματικών μας υπηρεσιών και αντιπροσωπιών ώστε να αναλάβει να τους υποδεχθεί. Η Νορβηγία ε, κάνει προσπάθεια για νέες εκλογές ελεύθερες, ανώθευτες και διαφανείς. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τις προσπάθειες που καταβάλλονται και από την πλευρά αυτή που επιδιώκει και ζήτησε πρόσφατα να εγκαταλείψουν την εξουσία αυτή που την έμονται παράνομα. Νομίζω ότι είναι λόγια τα οποία πρέπει πολύ γρήγορα, καθώς είναι λογικά λόγια, ε, σωστά λόγια, να υλοποιηθούν ταχύτατα. Ο επόμενος ομιλητής μας δεν βλέπω να είναι εδώ, λέει ο ομιλητής. Α, είσαστε εδώ μάλιστα. Και ευχαριστώ. Ο κύριος Νικόλαου Αλαβάνος Έχετε το λόγο για ένα λεπτό από τις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης της νέας δημοκρατίας ήταν να αναγνωρίσει τον αρχιπραξικοπηματία γκουαϊδό τον αχυράνθρωπο των ηνωμένων πολιτειών της αμερικής σαν μεταβατικό πρόεδρο της βενεζουέλας πατώντας ακριβώς πάνω στην απαράδεκτη κοινή θέση της ευρωπαϊκής ένωσης που στήριξε η κυβέρνηση του σύριζα. πρόκειται για πράξη που στηρίζει τη βρώμικη επέμβαση των ηνωμένων της ευρωπαϊκής ένωσης και των συμμάχων τους στη βενεζουέλα και στρέφεται κατά του νόμιμα εκλεγμένου προέδρου της χώρας και συνολικά κατά του βενεζουελάνικου λαού ο οποίο είναι ο μόνο υπεύθυνο για να καθορίσει τι πολιτικέ και κοινωνικέ εξελίξει στη χώρα του. ο ελληνικό λαό όπω πολλέ φορέ έχει κάνει στο παρελθόν χρειάζεται αποφασιστικά και τώρα να καταδικάσει την επέμβαση των ηνωμένων πολιτειών και τη ευρωπαϊκή ένωση στη βενεζουέλα μαζί και την αναγνώρισή τη από την κυβέρνηση τη νέα δημοκρατία που παίρνοντα τη σκητάλη από το ΣΥΡΙΖΑ παίζει το παιχνίδι των υπεριαλιστών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα εκφράζει τη διεθνιστική του αλληλεγγύη στο λαό τη Βενεζουέλα στο κομμουνιστικό του κόμμα και την κομμουνιστική νεολαία της χώρας που μάχονται για τα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστώ, Ντάβιτ Λέγκα. κύριε Υπατή εκπρόσωποι. Το σκαίο πρόσωπο του κομμουνισμού έχει πολλές μορφές και βλέπουμε στην Βενεζουέλα τον ε, Μαδούρο να έχει καταστρέψει τη χώρα αυτή που κάποτε ήταν τόσο πλούσια. Έχουμε ποσοστά μέχρι και 10 εκατομμύρια της εκατό ε, πληθωρισμού μέσα στην περίοδο στο 2019 πεινάει, ε, λιμοκτονεί ο κόσμος ενώ αν κατέβει στους δρόμους ε, βάλου ουραναντίον του οι δυνάμει του Μαδούρο. Είναι πολλά τα εκατομμύρια που έχουν φύγει από τη χώρα με βάση τα στοιχεία των ΗΕ. Οι Βενεζολάνοι έχουν γονατίσει, αλλά δεν έχουν ιτηθεί. Ο Χουάν ο Αϊδό είναι ο προσωρινό προσωρινός πρόεδρος τους, νομοποιημένος προσωρινός πρόεδρος τους, αναγνώριστηκε άλλωστε και από το Κοινοβούλιο και από τα περισσότερα κράτη-μέλη. Ωστόσο κάποια κράτη-μέλη εξακολουθούν να υποστηρίζουν ε, το παράνομο καθεστώς του Μαδούρου και με βάση αυτή την υποστήριξη συνεχίζονται τα εγκλήματα του καθεστώς του Μαδούρου ω ε, κατά του λαού τη Βενεζουέλα. Και γι' αυτό και θα τον γράψει με αυτούς τους όρους η ιστορία στα μελανά βιβλία. Πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική που προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στη Βενεζουέλα και ο Μαδούρο να κληθεί να δώσει λόγο για τα εγκλήματά του. Ευχαριστώ η κυρία Μπεάτα Κέμπα. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα γίνεται όλο και χειρότερη. Αν δείτε τις ενέργειες της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούμε ε, να βοηθήσουμε τους Βενεζολάνους όπως μπορούμε. Είναι προφανές ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά μόνο η διεθνής πίεση είναι αυτή που έχει φέρει την πλευρά του καθεστώτος στο τραπέζι των δραματεύσεων. Έχουμε δει βίντεο ε, με τους Βενεζολάνους και πόσο υποφέρουν. Έχουμε διαβάσει πως ε, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει, τι δεινά περνούν ε, ηλικιωμένοι παιδιά, γυναίκες ε, σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Και, αν, και παρότι προσπαθούμε να στείλουμε και τρόφιμα και φάρμακα, από την άλλη πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια πολιτική λύση Εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσουμε και του πολίτε και να δούμε οποιαδήποτε λύση, οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να παράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ ε, το λαό τη Βενεζουέλα. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και την άμεση αποστολή ε, βοήθεια στη χώρα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν όλοι ομιλητέ στον κατάλογο. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye. Πέντε λεπτά έχουμε στη διάθεσή μα. Και τέσσερι ομιλητέ. Πρώτη κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίτσια. Gracias. Κύριε Μπαραντικά, ευχαριστώ κύριε Μαγκερίνη. Τα συμπεράσματα των ΗΕ για την κατάσταση στη Βενεζουέλα κάνουν όλο και πιο πήγον να, να εργοποιηθεί μια ανθρωπιστική βοήθεια και μια μεταβατική διαδικασία προς τη δημοκρατία. Οι σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταστολή πρέπει να σταματήσουν. Ο σημερινό διάλογος έχει χάρτη πορεία σε δημοκρατικές ελεύθερες εκλογές και με συνθήκες για όλους με διεθνείς μηχανισμούς μηχανισμούς ε, που θα αποφύγουν την κατάχρηση της ε, λαϊκής βούλησης οι αριθμοί ε, των δολοφονηθέντων και των εξόριστων ουσιαστικά δικαιολογούν επέμβαση του ποινικού δικαστηρίου και επιβολή κυρώσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν οι Ευρωπαίοι πραγματικά νοιάζονταν για τους Βενεζολάνους, θα συγκεντρώναμε τρόφιμα και φάρμακα για εκείνους σε συνεργασία με την ε, ε, δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Μπορεί να μην συμπαθείτε το Μαδούρο, αλλά δημοκρατικά εξελέγει και υπάρχει υποχρέωση προς το λαό και για να ε, αντιπαλέψουμε τη βαναυσότητα των κυρώσεων ε, που πλήττουν τη Βενεζουέλα. Δεν έχουν κανένα νόημα αυτέ οι κυρώσει. Είναι μια νέα μορφή τρομοκρατία, γιατί στρέφονται κατά όσων πλήττονται περισσότερο και υποφέρουν περισσότερο. Θα ήταν καλύτερο μάλιστα ο Αμερικανικός στρατός να επέμβει, ε, να εισβάλλει στη χώρα και τουλάχιστον εκείνοι θα μπορούσαν να μηνθούν ε, νομίμω. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι χειρότερη μορφή οικονομικού πολέμου. Η απόφασή σας να στηρίξετε τον Κουαϊδό, έναν ακροδεξιό, ε, χωρίς καμία στήριξη, ήταν τεράστιο σφάλμα. Και λέτε ότι σας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο. Μα αυτό που κάνετε αντίκειται 100% στο διεθνές δίκαιο και οποιοδήποτε έχει γνώση των, της ένομης τάξης θα το επιβεβαιώσει. Πρόεδρε, είναι προφανές τώρα ότι η αναγνώριση του Γουαϊντό προσωρινού Προέδρου από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου όχι μόνο ήταν παράνομη η δύναμη του Βενεζολάνικου αλλά και του διεθνούς δικαίου. Ε, ταυτόχρονα όμως δεν έφερε και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το ότι κάποιοι βγαίνουν για να μιλήσουν για ανθρωπιστική καταστροφή όταν και για εκατομμύρια πρόσφυγες ενώ ταυτόχρονα προτείνουν στοχευμένα μέτρα και περισσότερες κυρώσεις, περισσότερα δεινά δηλαδή και, το λόγο, και περισσότερους λόγους για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τα σπίτια τους, πρέπει να πω ότι για μένα έχει ξεπεράσει και τα όρια ακόμα της υποκρισίας. Το να, μιλείτε, μιλάτε για ε, παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, ενώ έχετε μόλις κλείσει συμφωνία με την ε, Βραζιλία, της οποίας ο πρόεδρος έχει δώσει εντολή να πυροβολούν και να σκοτώνουν πολίτες στο δρόμο. Εάν σε απασχολούν τόσο ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί δεν κοιτάτε τα παγωμένα αυτά ε, οικονομικά ε, ε, στοιχεία ενεργητικού που είναι παγωμένα σε όλο τον κόσμο να απελευθερωθούν για να γυρίσουν πίσω στο λαό της Βενεζουέλας. Γιατί δεν κοιτάτε να δώσετε βοήθεια ανθρωπιστική, το να οδηγείτε στη λιμοκτονία ένα λαό ολόκληρο δεν έφερε ποτέ αποτέλεσμα, ούτε και πρόκειται εδώ να φέρει. Thank you, Mr. Ulrich Milan. Ευχαριστώ, Ulrich Milan. Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη. Κοίταξα το σχέδιο ψηφίσματος και άκουσα με προσοχή τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων και της δική σας. Μόνο όμως ε, κλισέ βλέπω να επαναλαμβάνονται και να αντικατοπτρίζεται η άβουλη αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει το παραμικρό. Μιλάτε για τη Βενεζουέλα, όπως άλλωστε και τη Λιβύη και, και στην περίπτωση της Λιβύης και του Ιράκ και του Ιράν. Αυτές οι καταστάσεις οφείλονται στην παρεμβατική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και τη στάση τους που με ένοπλη παρέμβαση δημιουργεί καταστροφές και τραγωδίες σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά για το χρήμα, για το πετρέλαιο. Αυτό δεν το λέτε στο σχέδιο ψηφίσματος, αγαπητοί συνάδελφοι. Ούτε λέξη γι' αυτό. Και γι' αυτό το ψήφισμα αυτό είναι τελείως χωρίς περιεχόμενο. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Έχουν εκπνεύσει τα πέντε λεπτά και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εφ' εξής, κατά τη διάρκεια της τρέχουσα θητεία θα τηρώ αυστηρά το πεντάλεπτο για, τις, ε, για τη διαδικασία γιατί αυτό προβλέπουν και οι διαδικασίες άλλωστε. Ακόμα και αν υπάρχει κάποιος ομιλητής ή ομιλήτρια που δεν γνώριζε ότι ε, υπήρχε το θέμα αυτό και καθώς κυρία Περέιρα δεν το γνώριζε ότι υπήρχαν αυτοί οι κανόνες θα της δώσω το λόγο κατ' εξαίρεση σήμερα αλλά θα την ε, παρακαλέσω από εδώ και μπρος να ξέρετε να λαμβάνετε υπόψη όλοι, όλοι ότι δεν θα ξεπερνάμε το πεντάλεπτο κυρία Περέιρα Ευχαριστώ. Βλέπουμε μια ε, υποκρισία και δημαγωγία αυτού του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει την επίθεσή της κατά της Βενεζουέλας και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ε, ε, ουσιαστικά επιμένετε σε συστηματικές δράσεις εσωτερικής αποσταθεροποίησης, τρομοκρατίας, σαμποτάζ, κυρώσεις, οικονομικό μπλοκάρισμα, διπλωματικό και χρηματοοικονομικό. Ε, όμως ε, ε, υπάρχει πολύ μεγάλη πορτογαλική ε, κοινότητα σε αυτή τη χώρα και την θέτεται σε κίνδυνο, όπως και τους πολίτες της Βενεζουέλας, υπερασπίζονται το διάλογο και την ειρήνη και υπερασπίζονται το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να αποφασίσει για το μέλλον του. Ε, αυτή είναι η λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Έχουμε έτσι ολοκληρώσει τον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρου των ε, βουλευτών και θα παρακαλέσω τώρα την ε, υπατή εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη Λόρο να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ποτέ ξανά δεν έχω ακούσει κάποιον ε, να εύχεται εδώ μία στρατιωτική επέμβαση. Και ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μου προκαλεί τρομερή έκπληξη και σοκ. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι που η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, προσπάθεια που καταβάλει, με το contact group, ε, μπορεί να διώξει σκέψεις ε, μια στρατιωτικής κλιμάκωσης είτε εντό είτε εκτός της χώρας. Είμαι περήφανη που εμείς είμαστε εκείνοι που εργάζονται μαζί με, τους, με τις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και, τους, και επιτρέπουμε σε εκείνους να μπουν στη χώρα και να παραδώσουν ε, τη βοήθεια αυτή. Είμαι περήφανη που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μεγαλύτερος ε, δωρητής λοιπόν, ε, ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα. Ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου και πραγματικά το ελπίζω, καθότι εμένα μόνο μερικοί μήνες μου μένουν ακόμα εδώ. Ελπίζω λοιπόν πραγματικά ότι εσείς θα αξιοποιήσετε τα επόμενα πέντε χρόνια χωρίς ε, να σκέφτεστε ότι είναι καλή λύση μια στρατιωτική εισβολή. Εμένα ως Ευρωπαία αυτό με τρομοκρατεί σαν σενάριο και αυτό θα πρέπει να ισχύει για οποιονδήποτε στην Ευρώπη. Γιατί εμείς έχουμε ζήσει στο πετσί μας τι σημαίνει ο πόλεμος και νομίζω ότι η αξία ε, του έργου μας είναι ακριβώς η ιστορία μας που είναι γεμάτη αίμα. Και αυτό μας έχει διδάξει ότι ο πόλεμος ποτέ δεν είναι καλή ιδέα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και νομίζω ότι υπάρχει σημαντική σύγκληση ε, στην Ολομέλεια, όχι ομοφωνία βέβαια, δεν περιμένει και κάτι τέτοιο, για την αναγκαιότητα να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρώτον, να βρούμε μια ειρηνική λύση Χωρί καμία στρατιωτική ε, απόπειρα. Δεύτερον, δημοκρατική λύση με, με εκλογές και όλες τι δικλείδε ασφαλεία, όλες τι διασφαλίσει ότι θα είναι ε, δίκαιες και ελεύθερες, που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Τρίτον, αυτό περιλαμβάνει δημοκρατικό διάλογο, πλήρη στήριξη είναι κάτι το οποίο κάνουμε και πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίε υπό την αιγίδα τη Νορβηγία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ξέρουμε, χωρί να είμαστε αφελεί, ότι και στο παρελθόν, με προηγούμενε τέτοιε απόπειρε, ε, τελικά είδαμε ότι δεν ήταν επιτυχή, ήταν πολύ δύσκολε και δεν απέφεραν καρπού. Όμω, θέλουμε ξεκάθαρη δομή, ξεκάθαρη προοπτική και νομίζω ότι είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου να υποστηρίξουμε αυτή την προοπτική μιας ε, δημοκρατικής ε, πολιτικής μετάβασης. Αυτό περιλαμβάνει και κυρώσεις. Και το ξεκαθαρίζω γιατί ελπίζω τουλάχιστον όσοι είστε εδώ σήμερα ξέρετε ποιες πολιτικές έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες όχι. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κυρώσεις κατά της χώρας ή του λαού της. Τα μέτρα που έχουμε υιοθετήσει στοχεύουν συγκεκριμένα μεμονωμένα άτομα που ευθύνονται για σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήθελα να είμαι απολύτω σαφή ω προ αυτό το σημείο. Τέλο, ανθρωπιστική βοήθεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε Πρώτο, πρώτα απ' όλα να παράσχουμε πόρους. Μίλησα με τη ΛΟΠΟΚ ε, προσφάτως, ε, αρμόδια για ζητήματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Μου είπε λοιπόν ότι σε αυτό το στάδιο, σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, το βασικό πρόβλημα λοιπόν είναι η έλλειψη πόρων και όχι τόσο η πρόσβαση. Ευθύνη μας λοιπόν είναι να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε τα επίπεδα βοήθειας προς ε, τους Βενεζολάνους, τα αδέρφια μας εκεί. Έχουμε τόσους δεσμούς. Έχουμε ακόμα και Βενεζολάνους εδώ μέσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μας να υποστηρίξουμε τον λαό της Βενεζουέλας. Αναμφίβολα. Όμως καθήκον και ευθύνη μας είναι να καλέσουμε και άλλους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια γιατί εργαζόμαστε φυσικά για την ε, διεξαγωγή δημοκρατικών και διαφανών εκλογών, παράλληλα όμως δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ε, δραματικές, ε, την δραματική ανθρωπιστική κατάσταση του λαού εκεί και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται και με την ενίσχυση ακόμα και των κυρώσεων και πάλι όμως κατά, μάλλον λαμβάνοντας στοχευμένα μέτρα. Ακολουθώντα τι πρόσφατε εκθέσει ε, για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι εξαιρετικά σοβαρέ. Ελπίζω λοιπόν, αν όχι όλοι, τουλάχιστον η μεγάλη πλειονότητά σα να μα υποστηρίξει σε αυτή την προσέγγιση. Γιατί ε, το να έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια ισχυρή φωνή εδώ, ε, είναι θεμελιώδου σημασία για να δραματίσουμε σημαντικό ρόλο από κοινού και με τι χώρε τη ευρύτερη περιοχή που συμμετέχουν στο Διεθνές Contact Group προκειμένου η Ευρώπη να αποτελέσει ε, τμήμα μιας ε, χρήσιμης και επικοδομητικής λύσης. Ευχαριστώ θερμά την Αντιπρόεδρο κυρία Μογκερίνη. Ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση. Σας ενημερώνω ότι έχουν κατευθεί έξι προτάσεις ψηφίσματος. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Πέμπτη. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και περνούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης δηλώσεις της ε, Αντιπρόεδρου για την κατάσταση του Περσικού κόλπου. Και παρακαλώ κυρία Μογκερίνη να πάρτε το λόγο για λίγο. φορά. Πρόεδρε ευχαριστώ. Ο Περσικός κόλπος είναι πολύ κοντά στην Ευρώπη. Έχουμε στενούς δεσμούς και έχει και στενούς δεσμούς και με τη δική μας την ασφάλεια. Έχουμε πει εξ αρχής ότι για μας είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα θέμα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Και αυτό το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Ούτε στρατιωτική ε, κλιμάκωση θέλουμε, ούτε αγώνα σε πυρηνικά όπλα. Έχουμε πει εξ αρχής ότι χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που είναι ήδη αρκετά περιπλοκή θα μπορούσε να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη, πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είναι τώρα. Το έχουμε πει. Τώρα βλέπουμε όλο και περισσότεροι να δέχονται τη διαπίστωση αυτή, ακόμη και κάποιοι που ήταν επιφυλακτικοί έως και πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τη συμφωνία με το Ιράν. Αντιλαμβάνονται λοιπόν τώρα ότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία. Αυτό ακούω να λένε στις συνομιλίες που έχω και οι περιφερειακοί ηγέτες ε, της περιοχής του Περσικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο και οι ηγέτες του Ιράκ, του Κουβέιτ που συνάντησα κατά την επίσκεψή μου στην περιοχή του προηγούμενου Σαββατοκύριακο ε, με τους οποίους μάλιστα συζήτησα το πώς μπορούμε να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση, ε, τι είδους πρωτοβουλίες υποστήριξης μπορούμε να αναπτύξουμε και να αναπτυχθούν από τα ίδια τα κράτη της περιοχής ώστε να υπάρξει μια καλύτερη ε, συνεννόηση και συναντήληψη μεταξύ των κρατών. Κανείς δεν λέει ότι επιδιώκει τον πόλεμο. Κανείς δεν προχωρεί σε δηλώσεις που να δείχνουν ότι υπάρχει πρόθεση πολέμου στην περιοχή αυτή ή και, πέρα, και έξω από αυτήν. Αλλά σε μια τέτοια περιοχή, σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, μπορεί να υπάρξουν λάθος υπολογισμοί, μπορεί κάποιοι λάθος υπολογισμοί να οδηγήσουν σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση και αντιπαράθεση. Γι' αυτό εμείς, Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούμε κάθε εμπλεκόμενο παράγοντα να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και να σκεφτεί με βάση την λογική τις κινήσεις του. Αυτό κάνουμε σε σχέση με την πυρηνική συμφωνία από τη μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ. Εχθές είχαμε και συζήτηση με τους Υπουργούς των Εξωτερικών των 28 κρατών μελών στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και τα 28 κράτη-μέλη σας βεβαιώ ε, δήλωσαν ομόφωνα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε από κοινού για τη διαφύλαξη της πυρηνικής ε, συμφωνίας, συμφωνίας για τα πυρηνικά ακόμα και υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες. Πρέπει να το πράξουμε αυτό, πρέπει να έχουμε Πρέπει να γνωρίσουμε ότι έχουμε την ευθύνη να το πράξουμε αυτό. Την κατάσταση τη γνωρίζετε. Ίσως ποτέ δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο σήμερα. 14 μήνε από την αποχώρηση τη μονομέρη των ΗΠΑ από τη συμφωνία, το Ιράν δήλωσε ότι σταδιακά θα μειώσει το βαθμό συμμόρφωσης στη συμφωνία αυτή. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας που παραμένει η αρμόδια και μόνη αρχή για την αξιολόγηση ε, τη συμμόρφωση του Ιράν επιβεβαιώνει ύστερα από ε, χρόνια όπου επιβεβαιώνει την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν τώρα ε, επιβεβαιώνει η Διεθνής Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας ότι το Ιράν συσσωρεύει περισσότερο εμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτά που βλέπουμε λοιπόν ανησυχούν με τους υπουργούς των εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας ε, εκδώσαμε μια κοινή διακήρυξη, μια κοινή δήλωση όπου καλούμε το Ιράν να επανέλθει στην συμμόρφωση της, ε, στη συμμόρφωση προς τη συμφωνία, πράγμα το οποίο συνέβαινε μόλις έως και πριν από μερικές μέρες ακόμη. Ε, εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μια απολύτως σαφής βούληση του Ιράν να επανέλθει στο πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά όσο περισσότερο περάσει ο χρόνος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να γυρίσει πίσω στην πλήρη συμμόρφωση στο Ιράν. Το μήνυμα που προσφέρουμε στο Ιράν λοιπόν είναι γυρίστε πίσω, δηλαδή κάντε αυτό που κάνατε μέχρι τώρα ε, με τη συμμόρφωση στη συμφωνία προς το συμφέρον το δικό μας, προς το συμφέρον των Ιρανών, προς το συμφέρον το συλλογικό και βεβαίως και αυτό άλλωστε ήταν και η ε, λογική βάση της οποίας συνήφθη αυτή η συμφωνία με το Ιράν, γιατί ξέραμε ότι τέτοιου είδους συμφωνίες είναι προς το συμφέρον όλων των μερών συλλογικά και προς το συμφέρον της συλλογική ειρήνης, επιτρέψτε να το διατυπώσω έτσι. Ταυτόχρονα εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μας με τα κράτη-μέλη ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να επιδιώξουμε τουλάχιστον να περιορίσουμε τις συνέπειες της μονομερούς απόφασης των ΗΕ για επανεπιβολή κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Τον Ιούνιο είχε συγκληθεί μια νέα σύνοδος ε, στη Βιέννη της ε, ε, Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας που επιβλέπει ε, τη συμμόρφωση με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και τη Γαλλία, ε, Βρετανία και Γερμανία παρόντες ε, όπου επιδιώξαμε και εξασφαλίσαμε κοινή προσέγγιση για τις δηλώσεις και τις δεσμεύσεις πλήρους συμμόρφωσης από κάθε πλευρά. Αυτή η κοινή επιτροπή λοιπόν στη συνεδρίασή της στη Βιέννη αποφάσισε ταυτόχρονα πως οι εμπειρογνώμονες θα συγκληθούν σύντομα θα συναντηθούν σύντομα για να συζητήσουν και άλλα ζητήματα όπως ζητήματα εξαγωγών ε, ε, είτε σε ουράνιο είτε σε βαρύ είδο του Ιράν προς άλλες χώρες. Δύσκολα ζητήματα. Την ίδια μέρα που συνεδριάζαμε στη Βιέννη, η Γαλλία, η Γερμανία και το Εμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν σε κάποια βήματα λειτουργικά σε σχέση με το Ιράν, σε συμφωνία την οποία επί καιρό επεξεργάζονταν, σε συνεργασία βέβαια και υποστήριξη και από τη δική μου την υπηρεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση με μέσα και εργαλεία που είναι πλέον λειτουργικά λοιπόν και μπορούν να προχωρήσουν στην πρώτη καταγραφή συναλλαγών ε, τυπικά και μάλιστα αμέσως ε, δήλωσαν ε, κάποια κράτη-μέλη, 7 περίπου, ότι πρόκειται να ενταχθούν στο μηχανισμό αυτό. Μέχρι σήμερα και άλλα έχουν δηλώσει πώς εξετάζουν τη δυνατότητα να μπουν στο μηχανισμό ΕΣΤΕΞ. E Είχαμε και άλλες συνομιλίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδεχομένω να ενδιαφέρονται για αυτές τις συναλλαγές γιατί η διαφύλαξη της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν δεν είναι προς συμφέρον μόνο της Ευρώπης. Είναι και άλλοι στον κόσμο που μοιράζονται τις ανησυχίες μας επί παραδείγματι τον κίνδυνο για έναν αγώνα δρόμου σε εξοπλισμούς και διπυρηνικούς στην περιοχή αυτή. Άρα λοιπόν η διαφύλαξη συμφωνία είναι ευθύνη δική μα, είναι προς το συμφέρον το δικό μας ναι, όντως, αλλά ταυτόχρονα και κοινή ευθύνη για κάθε ε, κράτο του, κόσμου, τη Ιφιλίου. Και θέλω για άλλη μια φορά να υπενθυμίσω ότι δεν είναι διμερής ή έστω πολυμερή ε, συμφωνία η εν λόγω συμφωνία είναι μία συμφωνία που έχει υιοθετηθεί ομόφωνα από την ε, Γενική Συνέλευση των ΕΕ με ψήφισμα. Έτσι λοιπόν, εμείς ως Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι θα ήταν ευχαιρής ο δρόμος, καθόλου ευχαιρής μάλιστα δεν είναι. Ε, ωστόσο αυτό που επιδιώκουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά και θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει όπως έδρασε, καταρχάς δεν θα υπήρχε η πυρηνική συμφωνία, δεν θα είχε συναυθεί ή δεύτερον δεν θα είχε επιβιώσει ως σήμερα. Και συνεχίζω λέγοντας ότι εάν ε, χαθεί αυτή η συμφωνία, μόνο βία, ε, κλιμάκωση, κινδύνους και εντάσεις μπορούμε να περιμένουμε στην περιοχή μας, Αλλά αυτό βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και αποδεικνύεται ότι έχουμε δίκιο. Αυτό που μας όμω δεν είναι να αποδείξουμε ότι έχουμε δίκιο, αλλά να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά για να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Κανείς νομίζω σήμερα δεν πρέπει να υποτιμά τον κίνδυνο μιας κλιμάκωσης στο κίνδυνο για όλους μας, τη Μέση Ανατολή, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Άρα προς το συλλογικό μας συμφέρον να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε ένα τέτοιο σενάριο, καθήκον δικό μας, δικό μας για όλων των Ευρωπαίων και πιστεύω ότι στέκουμε ενωμένοι. Είναι ακριβώς αυτό και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε για να διαφυλάξουμε τη συμφωνία, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε η φωνή της λογικής, θα εξακολουθήσουμε να το πράττουμε για τη δική μας την ασφάλεια, για την ειρήνη στην ταραγμένη αυτή περιοχή και επειδή γνωρίζουμε ότι ακριβώς όταν υπάρχει πρόβλημα είναι υποχρέωση να μείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας και συνεργασίας. Είναι απαραίτητο να επενδύουμε στις δημο... διπλωματικές οδούς για την επίλυση των προβλημάτων. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και πρώτη ομιλήτρια είναι η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την παρουσίαση της σημερινής κατάστασης στον κόλπο η οποία γίνεται όλο ένα και πιο προβληματική γίνεται το νευραλγικό σημείο στον κόσμο. Η ικανότητα του Ιράν να μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς αποτελεί μεγάλη απειλή για την ευρωπαϊκή οικονομία. και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους για να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κατάστασης. Κυρία Μογκερίνη, αναφερθήκατε στην κατάσταση και στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ενωμένη για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να πείσουμε το Ιράν να συνεχίσει να σέβεται τη συμφωνία ακόμη και μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θέλουμε να υπάρξουν νέες κυρώσεις, θέλουμε το Ιράν να συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίκουλα, τον Ίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπατή εκπρόσωπε, πράγματι το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράση αποτελεί ένα τεράστιο επίτευγμα και χρειάστηκε χρόνια διαπραγματεύσεων. Ένα τεράστιο επίτευγμα τη Διατλαντική Συμμαχία, που η νέα κυβέρνηση, τον είπα, αρνήθηκε δεν ε, είναι θετικό στο να ξυλώνουμε τα επιτέγματά μας ε, και το πολυμερές ε, σύστημα κανόνων ή να αμφισβητούμε διπλωματικές επιτυχίες. Η συμφωνία είναι κλειδί για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και για την παγκοσμία ειρήνη και ασφάλεια είναι προς το συμφέρον όλες τις διεθνούς κοινότητες και των ΙΠΑ, των Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ιράν. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε για να διατηρήσουμε τη συμφωνία και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε αυτά οικονομικά ωφέλη, ενώ θα υπενθυμίσουμε στους Ιρανούς εταίρους ότι πρέπει να σέβονται πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΙΠΑ έχει μεγάλο αντίκτυπο σε μια ιδιασταθή περιοχή. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να μείνει ενωμένη και σταθερή και να λάβει μια ξεκάθαρη θέση που θα υπερασπίζει το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος, η κυρία Λουαζό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κυρία Υπατή εκπρόσωπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη σύναψη της Συμφωνίας της Βιέννης. Από την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία, η ευθύνη της Ευρώπης είναι ακόμη μεγαλύτερη για να διατηρήσει αυτό το ουσιαστικό στοιχείο της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής για την διάδοση των πυρηνικών όπλων. Σήμερα είναι ανησυχητική η κατάσταση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιβάλει εκ νέου μονομερείς ε, κυρώσεις και εξοεδαφικές. Το Ιράν έχει ξεπεράσει το όριο που είχε τεθεί σε ό,τι αφορά τον εμπλουτισμό και την αποθήκευση του ουρανίου. Ο Περσικός κόλπος ε, γνωρίζει μια ενισχυτική ένταση. Ε, ουσιαστικά αυξάνεται ο κίνδυνος σύραξη στον κόλπο και τα συμφέροντα των πολιτών και των επιχειρήσεων απειλούνται απέναντι σε αυτή την έκτακτη ανάγκη. για συγκεκριμένα μέτρα προτείνεται προκειμένου να συνεισφέρουν στην αποκλιμάκωση και ποιες είναι οι προτάσεις σας προκειμένου το Instex να καταστεί πλήρως ε, επιχειρησιακό και με τη συμμετοχή και επιπλέον κρατών μελών. Η κυρία Νόημαν. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η συμφωνία του Ιράν, με το Ιράν για τα πυρηνικά ήταν μια μεγάλη επιτυχία διπλωματική μιας ανωμένης Ευρώπης. Και γυναίκες ήταν μπροστά στη διαπραγμάτευση στην πρώτη θέση, κυρία Μογκερίνη. στι τέσσερα χρόνια όμως μετά αυτό, η αυτή η μεγάλη επιτυχία κινδυνεύει. Κινδυνεύει λόγω των κινήσεων ως ανεύθυνου Πρόεδρου των ΗΠΑ. Κινδυνεύει διότι το καθεστώς του Ιράν έχει αρχίσει και πάλι να επιταχύνει τον εμπλουτισμό να αυξάνει μάλλον τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύει και γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική δεν είναι επαρκή για να αντισταθμίσει αυτήν την κλιμάκωση. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Περσικό που δούμε σήμερα εδώ δείχνουν πως μία θριαλίδα, μία μόνο θριαλίδα μπορεί να οδηγήσει σε μία κλιμάκωση που κανείς δεν επιθυμεί. Έτσι λοιπόν όλοι μας σήμερα αλλά και τις επόμενες εβδομάδες πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην κλιμακωθεί περισσότερο η κατάσταση αυτή σε μια περιοχή η οποία ήδη έχει καταστραφεί από τόσους πολέμους και γι' αυτό καλωσορίζουμε ως ομάδα των Πρασίνων τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου για επιδίωξη περαιτέρω λύσεων. Ναι, το Ιράν πρέπει να συνομιλήσει με τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, υποστηρίξει προτάσεις για περιφερειακή ε, συνέλευση, διάσκεψη στην οποία θα κάτσουν στο τραπέζι όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες για να επιδιώξουν μια λύση. Αλλά είμαστε και σαφείς, αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν οι σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αντιμετωπιστούν επίσης